κύριοι, παρακαλώ καθίστε στα έδρανά σα. Θα περάσουμε στην ψηφοφορία, στην εκλογή των κοσμητόρων. Και αυτή ηλεκτρονικά θα γίνει η εκλογή αυτή ως ψηφοφορία. Έχω τις εξή υποψηφιότητες που υπευλήθησαν. Έχουμε τους εξής υποψηφίους. Κάθριν Μπιέντα, Κορνέλιος Ντε Γιόγκ, Καρσκι, Ανδρέι Κόβατσεφ, Μπογουσλαβ Λιβεράτσκι και Elisabeth Morin Σαρκέ. Οι υποψήφιες, κυρίες και κύριοι, είπαν ότι με τη σύμφωνη γνώμη τους προτείνονται ως υποψήφοι. Υπενθυμίζω ότι στον πρώτο και δεύτερο γύρο απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία, στον τρίτο γύρο αρκεί η απλή πλειοψηφία. Η εκλογή θα γίνει όπως ακριβώς έγινε χθες ε, η εκλογή των αντιπροέδρων με τον ίδιο τρόπο. Έχουμε έξι υποψηφίους, γυναίκες και άνδρες για πέντε θέσεις, για πέντε αξιώματα. Θα είναι λοιπόν έγκυρα τα ψηφοδέλτια επί των οποίων το πολύ πέντε, πέντε όπου πέντε ονόματα θα αναφέρονται, πέντε υποψήφοι θα αναφέρονται. Δεν είσαστε υποχρεωμένοι να εκλέξετε πέντε, μπορείτε να εκλέξετε έναν ή παραπάνω από έναν, αλλά όχι πάνω από πέντε. Και ρωτώ τώρα γιατί τα τεχνικά θέματα. Απαιτείται κάποια αποσαφήνιση από πλευρά σας και πάλι. Ή μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η διαδικασία όπως χθες ε, ακολουθήθηκε είναι πλέον γνωστή σε όλους. Τουλάχιστον ο συνάδελφος Φεχόφστα το επιβεβαιώνει αυτό. Και μια και δεν βλέπω να υπάρχει κάποια ένσταση ή αντίρρηση, λέω και θεωρώ ότι μάλιστα αυτό έχει αφομοιωθεί, είναι πλέον γνωστό και έτσι θα γίνει. Ωραία λοιπόν και περνάμε τώρα στην εκλογή των κοσμητόρων κυρίες και κύριοι. Άρχεται η ψηφοφορία. haben Ψηφίσατε όλοι και όλες και όλοι, κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές. Ναι, also Moment Μια στιγμή, ακούστε. Μια στιγμούλα, τι συμβαίνει. Δεν αποφάσισα εγώ να γίνει αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι βρίσκονται στην αίθουσα και δεν είναι δυνατόν να κλείσει η ψηφοφορία χωρίς να έχει ολοκληρωθεί σωστά. Δεν γίνεται αυτό, εντάξει. Λοιπόν, δεν είχα πει πέρας ψηφοφορίας. Μπαίνουν διαρκώ στην αίθουσα και άλλοι συνάδελφοι. Πρέπει να ακυρωθεί η διαδικασία και να ξεκινήσουμε. Δεν είναι δυνατόν να γίνει έτσι όπως ε, έγινε. Κυρίες και κύριοι, μια στιγμή προσέξτε παρακαλώ. Δεν ξέρω τι συνέβη με τα τεχνικά, με τις συσκευέ και τους τεχνικούς, αλλά πιστεύω ότι δεν είπα ότι έληξε η ψηφοφορία. Εντάξει, και έτσι δεν μπορούμε να καταμετρήσουμε ψήφους επειδή είχαμε καταχωρήσει στη μία η ώρα την εκλογή αυτή, είναι τώρα μία και πέντε, πολλοί μπαίνουν στην ε, αίθουσα, οφείλεται και στα, στους ανελκυστήρες η καθυστέρηση. Δεν είπα ότι έληξε η ψηφοφορία, θα επαναλάβουμε λοιπόν την ψηφοφορία, εντάξει, παρακαλώ. Πρόεδρε, είναι μία ερμηνεία και θεωρώ, Πρόεδρε, ότι είναι προφανές όταν αρχίζει μια ψηφοφορία από τον Πρόεδρο καθορίζεται από το εκλογικό σώμα. Φυσικά στην Ολομέλεια υπάρχουν κάποιοι ευρωβουλευτές που μπαίνουν, κάποιοι άλλοι που βγαίνουν. Δεν μπορεί αυτό να είναι το κριτήριο για μια παράταση ψηφοφορίας. Μπαίνουν πάντα ευρωβουλευτές στην Ολομέλεια και πάντα συμβαίνει αυτό. Δεν μπορούμε λοιπόν να παρατείνουμε επαόριστο και γι' αυτό πρόεδρε ολοκλήρωσα, ολοκληρώνω να επαναλάβουμε την ψηφοφορία μπορεί να υπονομεύσει το αποτέλεσμα που επετεύχθη. Εξέφρασαν τη βούλησή τους οι ευρωβουλευτές, αποφάσισαν, ψήφισαν. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κανό, τους κανόνες του παιχνιδιού όταν το παιχνίδι είναι υπό εξέλιξη. Πρόεδρος, κύριε Ευρωβουλευτά, σε αυτό το σώμα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες και οι κανονισμοί. Ο κανόνας λέει ότι τότε θεωρείται ότι ολοκληρώνεται μια εκλογική αναμέτρηση όταν ο πρόεδρος λέγει ότι ολοκληρώθηκε. Εγώ δεν είπα ότι ολοκληρώθηκε η εκλογή. Αυτή την ψηφοφορία δεν είπα ότι ολοκληρώθηκα. Αν κάποιος τεχνικός σε αυτό το σώμα πατάει κάποιο κουμπί, δεν μπορώ εγώ να το αποφύγω, να οδηγήσω στο να αποφευθεί, αλλά αυτό δεν υπονομεύει την εκλογή, οπότε θα επαναλάβουμε τώρα την εκλογή. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για να πάνε όλα σωστά και να είναι όλα ορθά, και είναι μια θεμητή επισήμανση αυτή, αλλά για λόγους αλληλεγγύης με τους, για τους συναδέλφους που βρισκόντουσαν σαν ελκυστήρες και είχαν καθυστερήσει είπα ότι έπρεπε να αναμείνουμε τώρα λοιπόν θα αρχίσει η ψηφοφορία θα δώσουμε 2-3 λεπτά να ψηφίσετε και θα κλείσει η ψηφοφορία και όταν πω έληξε η ψηφοφορία μόνο τότε θα μπορέσουν οι τεχνικοί να πατήσουν τα κουμπιά για να καταμετρηθούν οι ψήφοι και παρακαλώ να το τηρήσουμε αυτό όπως προβλέπετε και όπως πρέπει λοιπόν κυρίες και κύριοι αρχίζει η εκλογή haben alle Abgeordneten Ψήφισαν όλοι οι ευρωβουλευτές. Dann ist der Wahlgang geschlossen. Τότε λοιπόν ολοκληρώνεται η διαδικασία. Λίγη εκλογή παρακαλώ να καταμετρηθούν ψήφοι. Das Ergebnis ist wie folgt. Το αποτέλεσμα έχει ω εξή. Κυρία Μωρά και 452 ψήφοι. Λιμπεράσκι, 443. Κύριε Μπέτρα, 425 ψήφοι. Κόβατσεφ 420 ψήφοι. Κάσκι 288, Ντε 152 ψήφοι. Η αναγκαία πλειοψηφία ήταν 339 ψήφοι. 677 ήταν οι έγκυρες ψήφοι. Εξελέγησαν λοιπόν η κυρία Μωράν Σαρτιέ, Λιμπεράτσκι, Μπίρντα και Κόβατσεφ. Συγχαρητήρια στην, για την εκλογή σας. Λοιπόν, χρειαζόμαστε και ένα δεύτερο γύρο στην εκλογή αυτή. Ερωτώ τους συναδέλφους Κάρσκι και Ντεγιόνγκ. Συμφωνούν, είναι υποψήφοι, εξακολουθούν και είναι υποψήφοι. Κύριε Ντεγιόν, τι λέτε. Ναι, εντάξει. Κύριε Κάρσκι, εσεί. Εντάξει, εξακολουθείτε και εσεί να είσαστε υποψήφιο. Παρακαλώ λοιπόν να περάσουμε σε αυτή την εκλογή. Άρχεται λοιπόν ο δεύτερος γύρος της εκλογής κοσμητόρων. Λογικά μία ψήφο μπορείτε να εκφράσετε. Πρέπει να αποφασίσετε υπέρ ποιου ε, υποψηφίου θα δώσετε αυτή την ψήφο που έχετε. Ψηφίσατε όλες και όλοι.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 Έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδικασίες για την εκλογή των κοσμητόρων. Συγχαίρω όλους που εξελέγησαν. Έχουμε μία ψηφοφορία τώρα για την αριθμητική σύνθεση των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Έχουμε την πρόταση της διάσκεψης των Προέδρων ως πρόταση. Όσοι είναι υπέρ να σηκώσουν το χέρι τους παρακαλώ αυτής της απόφασης. Υπέρ κατά αποχές